Παρακαλώ, λάβετε θέσεις. Ε, θα πρέπει να ξεκινήσουμε την ε, συνεδρίαση και την εκλογή. Έτσι. Σας καλωσορίζω λοιπόν ε, τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Είμαι ο Γιώσεφ Σάιερ, είμαι ο προσωρινός πρόεδρος της συνεδρίασης γιατί σύμφωνα με τον κανόνα, με το άρθρο 14, το μέλος που, είχε, που ήταν παρόν σε, για μεγαλύτερη χρονική περίοδο ε, προεδρεύει τη συνεδρίασης. Και ως εκ τούτου ε, δεν πρέπει να είστε γυρεός ε, για να λάβετε τη θέση του Προέδρου. Γιατί δεν μετράει η ηλικία, αλλά η υπηρεσία. Πόσο, ε, πόσο καιρό ε, έχω υπάρξει στην Επιτροπή. Παρότι λοιπόν έχω μουσια, δεν είμαι γυρεός. Θα ήθελα να επενθυμίσω ότι ότι ο σκοπός είναι να, να η σε συγκρότησε σώμα και να εκλέξουμε τον πρόεδρο σύμφωνα με τον κανονισμό 213. Ε, πρώτα θα εκλέξουμε τον πρόεδρο, μετά ε, ξεχωριστά τους αντιπροέδρους και σε περίπτωση που θα... Σας παρακαλώ λοιπόν, τα παρακαλώ τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη να έχουν τις κάρτες για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αν δεν την έχετε, μπορείτε να την ζητήσετε. Ε, αλλιώς θα πρέπει να κάνουμε ψηφοφορία σε χαρτί, η οποία θα είναι και πιο χρονοβόρα, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχουμε να εκλέξουμε ε, πολλούς υποψηφίους. Πρέπει λοιπόν να βρούμε όλη την ε, κάρτα μας. Θα σας δώσω λοιπόν το παράδειγμα. Λυπούμε, αλλά ήμουν... Ε, άφησα την κάρτα μου στο προηγούμενο, στο προηγούμενο, στην προηγούμενη αίθουσα ε, θα πρέπει να ζητήσετε ε, τον βοηθό σας λοιπόν να φέρει την κάρτα. Σε 10 λεπτά λοιπόν, ε, όσο το γίνεται το σημείο δυνατότερα να βρείτε την κάρτα σας παρακαλούμε. Τα ονόματα των αναπληρωματικών είναι τα ακόλουθα. Εύελιν Κέπχαρτ αντικαθιστά την κυρία Κατυπήρη που είναι πλήρες τακτικό μέλος. Σε αυτήν ε, είμαστε πολλά χρόνια λοιπόν στην Επιτροπή αυτή, αλλά ε, η διαφορά είναι ότι ενώ εγώ ήμουν τακτικό μέλος, εκείνη ήταν αναπληρωματική, ένα άλλο μέλος που ε, έρχεται ως εκπρόσωπος είναι ο κύριος Ανδρέα Καρόπο που αντικαθιστά τον κύριο Κολάρ, τακτικό μέλος ο κύριος Κολάρ, Εάν υπάρξει αλλαγή, τα πολιτικά, τα πολιτικά, οι πολιτικές ομάδες θα πρέπει να μας ενημερώσουν πριν την έναρξη της ψηφοφορίας. Ως προσωρινός πρόεδρος ε, θα προεδρεύσω ε, μόνο για την εκλογή του Προέδρου, μετά θα αναλάβει τα καθήκοντά του ο Πρόεδρος για την εκλογή των Αντιπρόεδρων. Αν υπάρχουν κάποια σχόλια, παρακαλώ. Όχι τότε προχωρούμε στην ε, ε, εκλογή του Πρόεδρου της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ε, υπάρχουν ε, φήμες ότι δεν έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες που τηρούνται εδώ και 40 χρόνια, δημιουργεί ένα μικρό θέμα σε εμά. Νομικά δεν ε, έχει κάποιο αντίκτυπο, αλλά ως Επιτροπή Νομικών Θεμάτων που εγγυάται την, το, το, το κράτος δικαίου και την καλή τήρηση των κανονισμών θα ήθελα να τηρούμε ε, τις παραδόσεις ε, των επιτροπών και των εκλογών και το του κράτους δικαίου φυσικά. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία, τότε έχουμε συνέπειες, ε, θα έχουμε συνέπειες για το μέλλον. Εδώ και 40 χρόνια ε, κινούμαστε με βάση αυτούς τους κανόνες, αλλά θα ήθελα λοιπόν να σας επενθυμίσω ε, την τήρηση των κανόνων εδώ. Προχωρούμε λοιπόν στην εκλογή του Προέδρου. υπάρχει απαρτία με το 1 τέταρτο των μελών, 7 μέλη δηλαδή, επομένως ε, ε, ζητάω, τον, ε, ζητάω τους συναδέλφους να μου πούνε τις υποψηφιότητες Ο κύριος Λεμπρετών. Σύμφωνα λοιπόν ε, ε, με το σύστημα στο οποίο αναφερθήκατε, έχω την τιμή να ε, προτείνουμε την υποψηφιότητα, προτείνουμε, αυτό προτείνουμε συγγνώμη για την Προεδρία. Είμαι μέλος της Επιτροπής εδώ και πέντε χρόνια. Ήμουν συντονιστής της ομάδας μου. Γνωρίζω πολύ καλά τα θέματα της ομάδας. Τα τελευταία πέντε χρόνια συμμετείχα στην, ε, σε, ε, σε πολλές ε, ψηφοφορίες, για, κυρίως για τα δικαιώματα του, του δημιουργού. Επίσης ήμουν εισηγητής για την άρση της ασυλίας, ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Είμαι καθηγητής δικαίου και επομένως θεωρώ ότι έχω όλα τα στοιχεία, όλα τα απαραίτητα προσόντα για αυτή την θέση. Υπάρχουν κάποια σχόλια. Επομένως, έχουμε μόνο αυτή την υποψηφιότητα. Να σας σταματήσω, δεν χρειάζεται να κάνετε σχόλια, απλώς ακούμε τις υποψηφιότητες ε, με βάση τους κανόνες. Ε, εκ μέρους του Renew Europe, η Lucy Φενσίγκερ είναι υποψήφια για την Προεδρία της Επιτροπής μας. Άλλος κανείς. Όταν έχουμε δύο υποψηφίους, πρέπει να ψηφίσουμε μυστική ψηφοφορία. Ζητώ από τους υποψήφιους να μας πούν αν δέχονται την ε, υποψηφιότητά τους. Για τον κύριο Λεμπρετό είναι σαφές. Αλλά για νομικούς λόγους θέλω να ακούσω ένα σαφές ναι ή όχι. Ναι. Και η άλλη υποψήφια δέχεται ε, την υποψηφιότητά της βεβαίως. Πολύ ωραία. Ε, πολύ ωραία. Έχουν ε, συμπληρώσει τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων και τη δήλωση ε, δέουσα συμπεριφοράς. Μέχρι στιγμής η συμπεριφορά σας είναι άψογη εντός της αίθουσας. Αλλά αυτό δεν είναι νομικά δεσμευτικό. Τα, οι υποψήφοι πρέπει να είναι τακτικά μέλη της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, το τσεκάραμε, ναι, και με βάση τον εσωτερικό κανονισμό το άρθρο 15.1 και το άρθρο 213, 3, έχουμε δύο υποψηφιότητες τις οποίες δεχόμαστε. Yes. I would like to remind that uh, I would like to remind that each member Κάθε μέλος που ψηφίζει έχει μόνο μία ψήφο με βάση την κατανομή των ψήφων στις πολιτικές ομάδες. 6 ε, το ΕΛΚ, 5 οι σοσιαλιστές, New Europe 4, πράσινοι έχουν 2. Το ID έχει 2, ECR έχει 2, GUE ένα ψήφο, μία ψήφο, συγγνώμη, και ράει ε, τρεις ψήφους. Συγγνώμη, οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Τρεις ψήφους. Πολύ ωραία. Έχετε, κυρία Γκέπχαρ, την κάρτα σας. Πολύ ωραία. Δεν έχουμε αλλαγέ ε, στα, στους αναπληρωτές. Η κυρία Γκέπχαρ, δηλαδή, είναι εδώ παρούσα και θα ψηφίσει. η εκλογή θα γίνει με απόλυτη πλειοψηφία. Θα δούμε ποιες είναι οι ψήφοι υπέρ του κάθε υποψήφιου. Αυτό θα δούμε μόνο. Και μπορείτε να ψηφίσετε μόνο υπέρ του ενός από τους δύο υποψηφίους. Το πράσινο κουμπάκι λέει ναι. Στο δεύτερο γύρο εκλέγεται ο υποψήφιος που έχει τις περισσότερες ψήφους. Ε, αν θέλετε να ψηφίσετε για τον κύριο Λεμπρετών, θα πρέπει να πατήσετε το πράσινο κουτί. Όσοι θέλετε να ψηφίσετε την κυρία Νάτσιγκα, θα πρέπει να πιέσετε το κόκκινο. Δεν μετράνε οι αποχές όταν υπολογίζουμε την πλειοψηφία. Φυσικά, εάν κάνετε λάθος, μπορείτε να αλλάξετε το κουμπί. Κάτι διάρκεια που τρέχει η ψηφοφορία. Αυτή τη στιγμή κλείσει η ψηφοφορία, δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία άλλη διόρθωση. Λοιπόν, αν είσαστε όλοι έτοιμοι, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε τώρα. more. Άλλοι δύο λείπουν που δεν ψήφισαν. So I close the vote. Πέρας προφορίας. 6. 23 ψήφοι έγκυροι. 16 υπέρ του κ. Λεμπρετών και 15 υπέρ της κυρίας Νέτσιγκα. κυρία Νέτσιγκα πήρε την, την απόλυτη πλειοψηφία. 15 και 6. 15 υπέρ της κυρίας Νέτσιγκα, 6 υπέρ του κυρίου Λεμπρετό, άρα εξελέγει η κυρία Νέτσιγκα. Σας δίνω το, τη θέση μου. Ευχαριστώ, συνάδελφοι, και χαίρομαι, είμαι πολύ ευγνώμων για την υποστήριξή σας. Και ελπίζω τα επόμενα πέντε έτη να επιτέλεσω το καθήκοντά μου στην Επιτροπή αυτή και να περάσουμε στις επόμενες ε, ψηφοφορίες ε, για την εκλογή των αντιπροέδρων. Έχουμε τέσσερις αντιπροέδρους. Θα ψηφίσουμε ξεχωριστά. Καταρχάς, για τον πρώτο αντιπρόεδρο, I would like to draw your attention to... Να σας επιστήσω την προσοχή στην πυκλομορφία ε, ε, του Κοινοβουλίου που θα πρέπει να αποτυπώνεται και στη σύνθεση του Προεδρείου. Θα πρέπει να έχουμε γυναίκες και άντρε και μάλιστα από πιο πολλά κράτη-μέλη. Για τη θέση λοιπόν του πρώτου αντιπρόεδρου έχουμε υποψηφιότητε. Σας ευχαριστώ. Ναι, θα ήθελα να υποβάλω την υποψηφιότητα του συναδέλφου μου Σεργέη Λαγκοντίνσκη. Ευχαριστώ. Άλλε υποψηφιότητες παρακαλώ. Ο κύριο Λεπρετό. Στο όνομα του πλουραλισμού θα υποβάλω και πάλι την υποψηφιότητά μου. Μάλιστα, θα γίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη θέση του πρώτου αντιπρόεδρου. the Λαγκοντίνσκι, πράσινο και κόκκινο κουμπί για τον κύριο Λεμπρετό. Έναρξη ψηφοφορίας, παρακαλώ. One more to vote. Μία ψήφος ακόμα, παρακαλώ. Πέρασε. Ο κύριος Λαμποντίνσκι εκλέχθησε. Συγχαρητήρια. And we will now move to the election και να περάσουμε στην ε, ψηφοφορία για τη θέση της δεύτερης αντιπροεδρίας. Η υποψηφία παρακαλώ. Ο κύριος Φως. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να προτείνω τον Μάριον Βάλτσμαν για τη θέση του δεύτερου αντιπρόεδρου. Μάλιστα. Άλλες υποψηφιότητε. Ο κύριος Λευριτό. Ναι, θα υποβάλω και πάλι την υποψηφιότητά μου στο πνεύμα, το προηγούμενο. Ε? Σας ευχαριστώ πολύ. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Η κυρία Βάλτσμαν, λοιπόν, ε, πράσινο και κύριος Λεμπρετών, ε, κόκκινο. Έναρξη ψηφοφορίας. Έναρξη ψηφοφορίας, πέρα ψηφοφορίας. Η ε, κυρία Βάλτσμαν, εξελεγείς. Ευχαριστούμε. Και συγχαρητήρια. Και τώρα περνάμε στην ψηφοφορία για τον τέταρτο αντιπρόεδρο. Τρίτο αντιπρόεδρο, δεν θα είναι πρόεδρος. Υποψηφιότητες, παρακαλώ. Καταρχάς, να σας συγχαρώ για την εκλογή σας στη θέση της Προέδρου. Συγχαρητήρια και καλή σας τύχη σας εύχομαι, γιατί είναι πολύ σημαντική η θέση εξ των σοσιαλιστών και με δημοκρατών. Τον κύριο Ντεμπλάνκο θα προτείνουμε για την θέση της, του τρίτου αντιπροέδρου. Άλλος παρακαλώ. Ο κύριος Λεπρετό. <laughs> Μάλιστα. Μα θα δοκιμάσω την τύχη μου τελευταία φορά, τρίτη και τυχερή. Ο κ. Γκαρσία Λαμπλάνκο συμφωνεί με την υποβολή τη υποψηφιότητά του, μάλιστα. Πολύ ωραία. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία, λοιπόν. Πράσινο για τον κύριο Γκαρσία Λαμπλάνκο και κόκκινο για τον κύριο Λεπρετού. Έναξη ψηφοφορία. Um, apologies, um, green... Ζητώ συγγνώμη. Πράσινο επαναλαμβάνει η πρόεδρο για την κυρία Κασίγια Μπλάνκο και κόκκινο για τον κύριο Λεμπρετό. Άλλοι δύο. Πέρασε. Ο κύριος Καρσία Ντελμπλάνκο εξελέγει. Και τώρα να περάσουμε στην ε, τέταρτη την Προεδρία. Υποψηφιότητες παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ ονόματος της ομάδος του ECR, ο κύριος Σταν Κανέλη, για την τέταρτη την Προεδρία. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς παρακαλώ. Όχι, αυτή τη φορά. Ευχαριστώ. Για να συνεχίσω στο πνεύμα των προηγούμενων εκλογών για την Αντιπροεδρία, θα ήθελα να ζητήσω η ψηφοφορία να γίνει μυστική. Πέντε μέλη πρέπει να ζητήσουν διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας. Μάλιστα, πέντε μέλη ζήτησαν μυστική ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά με μυστική ψηφοφορία, λοιπόν. να ελέγξω παρακαλώ αν ο κύριος Στανκανέλη συμφωνεί με την υποβολή της υποψηφιότητάς του, μάλιστα. Και μιας και έχουμε μόνο έναν υποψήφιο, θα ψηφίσετε, δεν έχουμε χρώματα, ή θα ψηφίσετε ή δεν θα ψηφίσετε. Πράσινο λοιπόν υπέρ, κόκκινο κατά. Έναρξη ψηφοφορίας. And we'll now close, close the vote. Thank you. Και έτσι λοιπόν ε, ε, εκλέγεται ο κύριος Στανκανέλη. So, I would like to give my... Να συγχαρώ λοιπόν όλους τους αντιπρόεδρους, να σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή σας. Έχουμε κάποια ανακοίνωση από πλευρά της Πρόεδρου. Επόμενη συνεδρίαση θα λάβει η χώρα στις 24 Ιουλίου. Σας ευχαριστώ. Πέρα στη συνεδρίαση.